Wir kommen jetzt zur Tagesordnung von... Äh, Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη της ΑΦΕΤ. Και εκεί επιζήτησε να συζητηθεί το θέμα της Τουρκίας. Θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε αύριο το απόγευμα. Νομίζω καλό είναι να συζητηθεί. Τώρα έχουμε... Α, δεν είναι εδώ η συνάδελφος. someone from the delegation to Moldova who has participated in that. Κάποιο από την αντιπροσωπεία τη Μολδαβία υπάρχει, ο κύριο Σόλτ ήρθε. Μάλιστα, μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στο επόμενο θέμα. Η ενημέρωση για τι ε, προεδρικέ εκλογέ Μολδαβίας. Κύριε Σόλτ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε να σας ενημερώσω για το ταξίδι της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προεδρικές εκλογές της Μολδαβίας. Είναι οι πρώτες άμεσες εκλογές Προέδρου της χώρας από το 1996. Όπως ξέρετε, αρκετοί από εσάς, είναι ο πρώτος γύρος μόνο ο πρόεδρος ε, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Ίγκορ που θεωρείται γενικά ρωσόφιλος, ε, έλαβε 48,5% και άρα ε, θα, πάει, θα πάνε σε δεύτερο γύρο. Κατόπιν δεύτερη ήρθε η κυρία Μαϊάσαντου, φίλο Ευρωπαία, με 38,2%. Η προσέλευση ήταν γύρω στο 50% των ψηφοφόρων. Βεβαίω η Μολδαβία πάρα πολύ ψηλά στα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο μας και βεβαίως συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις στην χώρα. Είχαμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε αυτό το μήνυμα και στις διμερείς επαφές μας με τον ε, πρόεδρο και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε, ήμασταν τμήμα μιας διεθνούς αποστολής παρατηρήσεων των εκλογών με άλλες και βεβαίως συντάξαμε από κοινού ένα σχέδιο δήλωσης το οποίο παρουσιάσαμε σε μια συνέντευξη τύπου και συμφωνήσαμε πλήρως με τα ευρήματά του. Και βεβαίως είχαμε, όπως είπαμε, την μικρή κοινοβουλευτική συνέλευση στο Κισνόβιον. Μπορείτε εκεί πέρα λοιπόν να δείτε τα περιεχόμενα της ανακοινώσή μας και καταλήξαμε στο ότι έγιναν σεβαστές οι θεμελιώδεις ελευθερίες και υπήρχε ανταγωνισμός στην προεκλογική εκστρατεία, όμως υπήρξε κάποια κατάχρηση διοικητικών πόρων, δεν υπήρχε διαφάνεια στα οικονομικά της εκστρατείας και δεν ήταν ισορροπημένη η κάλυψη των ΜΜΕ. Επανέλθω λοιπόν σε αυτά. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν την γενικά άψογη συνεργασία, οργάνωση της διαδικασίας και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων στα εκλογικά τμήματα. Στα τμήματα τα οποία ευσχεστήκαμε τρία τέταρτα των επιτροπών ήταν γυναίκες και είναι και δικό τους κατόρθωμα αυτό. Σε γενικές γραμμές λοιπόν ικανοποιηθήκαμε για το ότι είδαμε και πολλές γυναίκες ε, υποψηφίους. Τέσσερις από τις εννέα ήταν γυναίκες και όπως είπαμε μία από αυτές Επέρασε στο δεύτερο γύρο. Κάτι το οποίο είναι σαφής βελτίωση σε σχέση με το 2014. Νομίζω λοιπόν πως ε, πρόκειται για ένα σημείο καμπής για την Μολδαβία του μέλλοντος όπου όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτική ζωή και να ε, ανταγωνίζονται για τα δημόσια αξιώματα τόνισα επίσης ε, την ανάγκη τα ΜΜΕ να μην προωθούν στερεότυπα με βάση το φύλλο και να σέβονται όλους τους υποψηφίους. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, προσπάθειες να βελτιωθεί το πολιτικό κλίμα. Επίσης ε, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με διάφορους ενδιαφερόμενους, ΜΚΟ, ΜΜΕ και από κοινού με άλλους ε, αναφερθήκαμε στις βασικές μας ανησυχίες. Ε, το ένα είναι τα οικονομικά, η έλλειψη διαφάνειας ε, καθώς επίσης ε, και η δυνατότητα χειραγώγησης των μέσων που υπάρχει έτσι. Στις ε, προπαρασκευαστικές ε, συναντήσεις μας συζητήθηκε το θέμα της κάλυψης της προεκλογικής εκστρατείας και εξ ονόματος της αντιπροσωπείας μας πρότεινα και στα ΜΜΕ να δρουν σύμφωνα με κάποιους κανόνες ακαιρεότητας και να υπάρχει μια ισορμένη κάλυψη των εκλογών. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να μην υπάρχει διχαστική ρητορία και θα πρέπει ο λαός της Μολαβίας να ψηφίζει με βάση το πρόγραμμα των δύο Αναμένουμε λοιπόν τον δεύτερο γύρο στη, την Κυριακή ...13 Νοεμβρίου και βέβαια αναμένουμε τα αποτελέσματα της πρώτης άμεσης ψηφοφορίας για πρόεδρο της Μολδαβίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσατε και για την προσοχή σας. Äh, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, μέλος της αντιπροσωπείας παρατηρήσεις των εκλογών στη Μολδαβία με επικεφαλής τον κύριο Σόλτες θα ήθελα από τα εξής. Πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι συμφωνώ με όλα αυτά που είπε ο Ιγκο Σόλτους προηγουμένως. Είδαμε να είναι αμερόληπτες και ελεύθερες εκλογές στην ε, Μολδαβία. Είδαμε και στην πρωτεύουσα και στις επαρχίες την εκλογική διαδικασία. Στην πρωτεύουσα πρέπει να πω όλα τα μέλη των τοπικών εκλογικών επιτροπών ήταν πολύ καλά προετοιμασμένα, γνωρίζαν την νομοθεσία, ήταν ιδιαίτερα προδραστικά και οι εκλογές οργανώθηκαν με πολύ σωστό και επαγγελματικό τρόπο. Στις επαρχίες και εκεί ήταν σωστά οργανωμένη η εκλογική διαδικασία, αλλά είδαμε στην περιοχή του ΟΧΕΙ, όταν ο Δήμαρχος εκεί ποικοτάζησε τις εκλογές γιατί δεν έγινε δεκτός ο υποψήφιος που προτάθηκε από αυτούς, είδαμε να εμποδίσονται κάποιοι να ψηφίσουν. Αυτό αναφέρθηκε όμως στην αστυνομία και η αστυνομία επανέφερε την τάξη και αυτοί θέλαν να ψηφίσουν, τελικά μπόρεσαν όλοι να ψηφίσουν. Δεν υπήρξε λοιπόν νοθεία, δεν υπήρξαν ε, ατασταλίες, αλλά είδαμε να υπάρχει κάποια διαδικασία εκφοβισμού και εμποδισμού των ψηφοφόρων. Είμαστε επίσης και πολύ κοντά στα σύνορα με την υπερπνιστερία. Δεν είδαμε νοθεία, είδαμε όμως κάποιες εντάσεις. Είδαμε αναφέρθηκε ότι κάποιοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία και πούλμαν για να ψηφίσουν. Αυτό βέβαια δεν είναι παράνομο, αλλά φυσικά τους φέρανε για να ψηφίσουν υπέρ κάποιου συγκεκριμένου υποψηφίου. Λειτουργήσε πολύ καλά και το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και αυτό απέτρεψε την πολλαπλή ψηφοφορία και τις νοθείες, αλλά στην επαρχία, στην Ήπεθρο, είδαμε να υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Όπως είπε και ο Ιγκορ προηγουμένως, η αντικειμενική στάση των μέσων ενημέρωσης και η εκστρατεία των πολιτικών κομμάτων και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά ως τμήμα των σχέσεων που έχουμε με τη δημοκρατία της Μολδαβίας. Τα σημαντικά θέματα σε αυτή την εκστρατεία και τα οποία θα παραμείνουν μετά και τις εκλογές είναι ο αγώνας κατά της διαφθοράς, η ενίσχυση της δικαστικής εξουσίας, και να μπορέσει να διαλευκανθεί η απάτη αυτή που αφαίρεσε ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες. Όλα αυτά τα θέματα θα είναι και στο θεματολόγιο της επόμενης Προεδρίας στη Μολδαβία. Θέλω λοιπόν να υποστηρίξω όλα αυτά που είπε ο Ιγκο εν κατακλείδη και τον ευχαριστώ για τον πολύ σωστό και διάφορο τρόπο με τον οποίο <clears throat> ηγήθηκε τις αντιπροσωπείες μας και σύμφωνα με αυτά που είπε ότι ήταν ελεύθερες, αμερόληπτες και δημοκρατικές εκλογές και θα είμαστε πάλι παρόντες στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Κύριος Κριστέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυβέρνηση της, Μολδοβα, της Μολδαβίας για την πολύ καλή αυτή ε, διοργάνωση των εκλογών. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι προεδρική δημοκρατία η ε, Μολδοβία. Είναι σημαντικά τα αξιώματα του Πρόεδρου σίγουρα, αλλά περιορισμένα. Η κυβέρνηση είναι αυτή που καλείται να προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις, να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις. Αυτός μην το ξεχνάμε. Από όσο κατάλαβα, μέσα σε μερικές ώρες ενδεχομένως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μας δώσει κάποια θετικά νέα, εγκρίνοντας την συμφωνία που υπάρχει σε επίπεδο προσωπικού μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Μολδαβίας. Και τρίτον, να ευχηθώ καλή τύχη για την Μάια Σάντου, την υποψήφια που ανήκει στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσει με επικοδομητικό τρόπο το εκλογικό σώμα γνωρίζοντα ότι ε, ορισμένοι ψηφοφόροι του ε, Δημοκρατικού Κόμματος στη Μολτοβία είναι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε ρωσικά. Αυτό θα πρέπει να το έχει κατά νου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι όντως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το πλαίσιο στο οποίο εξελίχθηκαν οι εκλογές ήταν διαφανές και δημοκρατικό. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα πρόοδου και αποτελεί συμβολική ένδειξη των μεταρρυθμίσεων που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στα πλαίσια των πολιτικών που ακολουθεί η χώρα αυτή. Το νομικό πλαίσιο έχει ε, τροποποιηθεί όντως στην Μολδαβία. Αυτό υπόθηκε πολύ σωστά και από τους προλύσαντες. Και όντως πλέον ο πρόεδρος εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, αλλά εξακολουθεί να έχει περιορισμένες αρμοδιότητες στη χώρα αυτή. Μόλον ακούσαμε λοιπόν πάρα πολλές υποσχέσεις, και κάποιε αναφορές σε σκάνδαλα όσον αφορά την προεκλογική εκστρατεία, ας είμαστε κι εμείς λίγο ρεαλιστές και α συνειδητοποιήσουμε ότι οι εκλογέ αυτές μπορεί τελικά να μην επιφέρουν τεράστιες αλλαγέ. Πολλοί ήταν υποψήφοι για τις προεδρικέ εκλογές, πολλοί όμως παρετήθηκαν τελευταία στιγμή και νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει τελικά ότι επικράτησε η κοινή λογική ανάμεσα στους διάφορους υποψήφιους από τα διάφορα πολιτικά κόμματα. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Κριστέα πριν από λίγο, που συνεχάρει την υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λεκού Κόμματος, που συμμετέχει βέβαια ή θα συμμετάσχει στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Και αυτό όμως καταδεικνύει ότι τα πράγματα κινήθηκαν θετικά. Υπήρχε τώρα μία αρκετά έντονη ατμόσφαιρα όσον αφορά την εκλογική εκστρατεία. Ο Ίγκορ ο οποίος υπήρξε ο σημαντικότερος διαπραγματευτής για την ε, Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα έρχεται και λέει ότι θέλει να αναθεωρήσει τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Μολδαβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται πολύ συχνά στην ε, εγκαθίδρυση πιο στενών σχέσεων με τη Ρωσία. Τα πράγματα αυτά δεν συνάδουν όμω, δεν συνδυάζεται το ένα με το άλλο και από ό,τι φαίνεται ορισμένοι ψηφοφόροι στη Μολδαβία όντως εντυπωσιάστηκαν από τις υποσχέσεις του και τα μεγαλεπίβολα λόγια του και γι' αυτόν τον λόγο τον ψήφισαν. Εναπόκειται σε κάθε περίπτωση βέβαια στους πολίτες της Μολδαβίας να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρό τους Πιστεύω ότι ο επόμενος πρόεδρος θα καταφέρει να προχωρήσει περισσότερο με τις μεταρρυθμίσεις. Χρειαζόμαστε όλο και περισσότερες μεταρρυθμίσεις στην χώρα αυτή και ελπίζω ότι ε, δεν θα ακολουθηθεί αναγκαστικά αυτή ε, η ατζέντα κοινωνικής οικονομικής πολιτικής που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της προκλογική εκστρατείας είναι πολύ σημαντικό ο επόμενος πρόεδρος να εργαστεί για το μέλλον της χώρας και όχι εναντίον του οικονομικού μέλλοντος της χώρας αυτής. Έχουμε λοιπόν μία υποψήφια, την Μάια Σάντου, η οποία είναι, έχει υιοθετήσει προφανώς μια υποψηφια την μαια σαντου η οποια στάση και μιλάει και περισσότερο για το ευρωπαϊκό μέλλον της Μολδαβίας. Προφανώς λοιπόν την υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κύριος Καστάλντο. Μπορούσα και εγώ να συμμετάσχω σε αυτή την πολύ σημαντική αποστολή επιτήρηση των εκλογών. Θα ήθελα λοιπόν καταρχά να ευχαριστήσω το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διαθεσιμότητά του και τον επαγγελματισμό του. Και θα ήθελα όλο ιδιαίτερω να ευχαριστήσω βέβαια και τον επικεφαλή τη αποστολή αυτή, τον κύριο Ίγκορ Σόλτε, ο οποίο έκανε μια εξαιρετική εργασία, συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά με όλα τα μέλη τη ε, αποστολή αυτή. Και καταφέραμε όλοι κατά αυτόν τον τρόπο να εργαστούμε πικοδομητικά για την διεξαγωγή αυτής της αποστολής. Θα μπορούσαμε όντως να πούμε ότι η έκβαση της εκλογικής διαδικασίας ήταν θετική. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, η εκλογική νομοθεσία τηρήθηκε, δεν υπήρξαν ατασταλίες και παρατυπίες. Όπως είπε και ο προλαλής Όντως υπήρξαν κάποιες παρατυπίες μεμονωμένες, οι οποίες όμως στο σύνολό τους δεν επηρεάζουν την θετική έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Θεωρώ λοιπόν ότι όντως έχει σημειωθεί πρόοδος, αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε και να το αναγνωρίσουμε. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται στην κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κάποιος διχασμός. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε εμεί περισσότερο τη συνεργασία με μια χώρα η οποία θα πρέπει να κινηθεί περισσότερο προς τον ευρωπαϊκό δρόμο. Προφανώς ε, κάποια σκάνδαλα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα αυτή, κυρίως ε, το ένα αυτό δισεκατομμύριο δολάριο που εξαφανίστηκε από τις ε, τρεις σημαντικότερες τράπεζες της χώρας, ακόμα εξελίσσονται έρευνες για το σκάνδαλο αυτό το χρηματοοικονομικό και σε επαφές που είχαμε και με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και άλλους ηθήνοντες αλλά και με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της χώρας μας είπαν ότι όντως αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, τις ευθύνες τους προκειμένου να ολοκληρώσουν την έρευνα αυτή που έχει ξεκινήσει για, για το οικονομικό αυτό σκάνδαλο. Κατά τη διάρκεια μάλιστα τη αποστολή επέμεινε στο σημείο αυτό και ο κύριο Σόλτο, λέγοντα ότι θα πρέπει να γίνονται πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι και μετά τις εκλογές όσον αφορά τα οικονομικά της χώρας. Να τονίσω και κάτι ακόμα. Οι εκλογές αυτές γίνονται όπως ακούσαμε με καθολική ψηφοφορία. Το Σταγματικό δικαστήριο της χώρας αναγνώρισε παράνομο, παράνομη μία τροποποίηση η οποία ε, προσπάθησε να λάβει χώρα από κάποιους πολιτικούς στο παρελθόν, αλλά στη συνέχεια αναγνώρισε τη δυνατότητα εκλογής του Προέδρου με καθολική ψηφοφορία. Ας μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια τη προκλογική εκστρατεία αναφερθήκαν οι υποψήφοι πάρα πολλικές μεταρρυθμίσεις αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Κανονικά τα ζητήματα αυτά δεν άπτονται την αρμοδιοτήτων ενός Προέδρου σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η σχέση που θα δημιουργηθεί στο μέλλον ανάμεσα στον πρόεδρο αυτό, ο οποίος πλέον εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της χώρας και, από τον επικεφ... και σε σχέση με τον επικεφαλής της κυβέρνησης, με τον πρωθυπουργό δηλαδή. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε και κατά τον δεύτερο γύρο των εκλογών και κυρίως μετά τις εκλογές ποια θα είναι η σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά αξιώματα. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε αυτό και με τους συναδέλφους να καταφέρουν οι θύνοντες στη χώρα αυτή να εμείνουν σε κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρίως να υπάρχει διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί και ίδια η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετέθη ένα αμφιβόλο από ορισμένα κόμματα της χώρας αυτής, οι οποία δεν λειτουργήσαν με τον δέοντα τρόπο κάθε φορά που συνεργάζονταν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά πολλές φορές παρουσίασαν και κατά τη διάρκεια της προκλικής εκστρατείας την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μη αξιόπιστο εταίρο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε ότι όντω θα υπάρχει δέουσα σοβαρότητα από όλου του πολιτικού τη χώρα και μετά τις εκλογές και ιδίως τη στάση που διατηρούν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ικανοποιούμαι από το γεγονός ότι οι συναδελφοί μου αναγνωρίζουν ένα αποτέλεσμα το οποίο επετεύχθη δημοκρατικά ακόμα και αν δεν ήταν υπέρ του υποψηφίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε αποσύσει μεγάλες ε, αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν θα μπορούσαμε να είχαμε μάλλον αποτρέψει αντιπαραθέσει του ίδιου, του είδου αυτού, αυτού που έγινε στην Ουκρανία, αν είχαμε ακολουθήσει και εκεί αυτή την πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει μια πολιτική δημιουργία γεφυρών για να επιτρέψει μια ολοκλήρωση σε όλο το μήκο και το πλάτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και θα έπρεπε να αναγνωρίσει ότι μέσα στα πλαίσια αυτή τη πολιτική ολοκλήρωση θα πρέπει να είναι εταίρο μα και η Ρωσία. Χαίρομαι λοιπόν <clears throat> που ακούω ότι αναγνωρίστηκε το δημοκρατικό αποτέλεσμα των εκλογών και ότι θέλουμε κι εμείς να συμβάλλουμε να υποστηρίξουμε την ειρήνη και όχι τον πόλεμο στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ο πρώτος, ο πρώτος χωρίς μικρόφωνο, μια εκλογική επιτροπή παρακολούθησης έχει δι, έχει διακριβώσει ότι και στην περίπτωση της Ουκρανίας οι εκλογές ήταν ε, ελεύθερες και αμερόληπτες. Επομένως αυτό δεν πρέπει να το διαμφισβητήσει κανείς ούτε εσείς, είναι κάτι το οποίο είναι σαφές. Και εμείς από την πλευρά μας έχουμε τονίσει ότι ακόμα και στην ε, Κρυμαία υπήρχε μια, μια πλειοψηφία υπέρ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η θέλησή της παραβιάστηκε. Εμείς γνωρίζουμε βέβαια ότι ο κύριος Πούτιν βρίσκεται σε, θέση υποστήριξης προς την κυρία Λεπέν και το κόμμα της. Η κυρία Καλνιέται τώρα έχει να θέλει να λόγο. Σάνδρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι οι προεδρικές εκλογές στην Μολδαβία, ο πρώτος γύρος των εκλογών αυτών ήταν πράγματι ελεύθερες και δημοκρατικές. Θα ήθελα όμως να φέρω στην προσοχή των συναδέλφων και το γεγονός ότι θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος. Και υπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα στα οποία θα πρέπει να σταθούμε και να δώσουμε την προσοχή μας και να ευστιάσουμε και την προσοχή των Εθνικών Αρχών και της Εκλογικής Επιτροπής στα θέματα αυτά. Ένα από αυτά είναι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Αν το 80% των μέσων ενημέρωσης είναι υπό την εξουσία ενός ατόμου και μόνο, φυσικά αυτό θα επηρεάσει τα αποτελέσματα των εκλογών. Επίσης είναι γνωστό ότι στη Μολδαβία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο χρησιμοποιούνται διοικητικοί πόροι από την τοπική δηλαδή και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, πόροι που χρησιμοποιούνται από τις υποψηφίου οι οποίοι είναι δήμαρχοι ή εκεί. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξεταστεί και το θέμα της χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας. Υπάρχουν επίσης κάποιες ανισότητες και θα πρέπει η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή να αποδώσει μεγαλύτερη προσοχή σε, στην εφαρμογή του εκλογικού δικαίου σε όλη την επικράτεια της Μολδαβίας. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι ιδιαίτερα επισφαλές. Υπάρχουν πολλοί πολίτες της Μολδαβίας οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, ζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό. Ποια είναι η δυνατότητα να ψηφίσουν που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι μεγάλο ο αριθμό του. Και το τελευταίο σημείο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσω και το οποίο και αυτό είναι επίμαχο, είναι ο... η αλλαγή στον εκλογικό νόμο, το άρθρο 47, που απαγορεύει στα κόμματα να αναφερθούν σε πολιτικά σημαντικές προσωπικότητες. Μα ακόμα και χώρες της Αφρικής, οι οποίες δεν διεκδικούν το χρήσμα της δημοκρατίας, δεν έχουν τέτοιου είδους νομοθεσία. Θα ήθελα λοιπόν, μετά το δεύτερο γύρο, να μπορέσουμε να επανέλθουμε, να έχουμε τη δυνατότητα φυσικά να πούμε ότι ήταν αμερόληπτες και ελεύθερες εκλογές, αλλά να γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ομαλοποιηθεί η πολιτική κατάσταση στη Μολδαβία. Ευχαριστώ. I, I can tell you that if uh, Mr. was allowed... Κοιτάξτε, αν επιτρεπόταν στον κύριο Ντόντον να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τον κύριο Πούτιν, δεν θα έπαιρνε 60-70% θα έπαιρνε στη Μολδαβία. Αλλά ευτυχώς δεν το επιτρέπεται να κάνει κάτι τέτοιο. Erstens, wer lässt es nicht zu? Und zweitens habe ich es dennoch nicht verstanden. Πρώτον, δε, εντάξει, δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιο ζήτημα και δεύτερον, δεν, κατάλαβα. Ούτω ή άλλω τελειώσαμε με αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη και περνάμε στο επόμενο ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ζωτουή για το θέμα του υπερπολισμού τη αποστολή στην Γάζα. Τη αποστολή τη Επιτροπή του Υπερπολισμού στη Γάζα, μα Oh, to survive. Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο θέμα αυτό της ημερήσιας ε, διάταξης. Έχουμε εδώ πέρα τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού, ο οποίος επισκέφθηκε στην Λωρίδα της Γάζας ε, κατόπιν εντολής του Προέδρου Σούλτς που είχε δοθεί και σε μένα αλλά για διάφορους λόγους δεν μπόρεσα δυστυχώς να συνταξιδεύσω και ότι συνδύασε με ένα άλλο ταξίδι και πήγε στην Δυτική Όχθη και στη Γάζα για να δει πώς πηγαίνουν τα πράγματα, να δει και την ε, ανθρωπιστική κατάσταση και τον αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Οπότε, μέχρι να ταξιδέψει ο κύριος Σαρτουή κανείς ευρωβουλευτής δεν είχε λάβει άδεια να επισκεφθεί την Λόριδα της Γάζας από το 2011. Τώρα επιτέλους έληξε αυτό και Ελπίζω, κύριε συνάδελφε, να μην έχετε μόνο άσχημα νέα. Έχετε τον λόγο. Merci. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι που με δίνετε δυνατότητα να πάρω το λόγο σήμερα προκειμένου να κάνω ένα απολογισμό της ε, Αποστολή αυτής από τις 18-21 Ιουλίου 2016 τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στην ε, Δυτική Όχθη. Μετά από αίτημα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτ, έλαβα εντολή για να, κάνω, να πάω στην αποστολή αυτή ως πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών, με απότερο στόχο να καταφέρω να αποτιμήσω την χρήση των κοινοτικών κονδυλίων που γίνεται επί τόπου κονδύλια τα οποία αποστέλει προς την Παλαιστίνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. 300 περίπου εκατομμύρια τα οποία δίδονται κάθε χρόνο στην Παλαιστίνη και τα οποία κάνουν τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση τον πρώτο και σημαντικότερο χρηματοδότη της περιοχής αυτής. Θα μπορούσαμε αγαπητές συνάδελφοι να είχαμε πάει μαζί σε μια κοινή αποστολή με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, δυστυχώ όμω δεν μα το επέτρεπαν οι ενηλυμένε μα υποχρεώσει, όπω είπατε. Και ω βασική προπόθεση είχα θέσει το εξή. Όπω το είπατε κι εσεί, κανένα Ευρωβουλευτή δεν είχε πάει στη Γάζα από το 2011 και μετά. Και λαμβάνοντα υπόψη τις οδηγίες που μου δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Μπόρεσα να περάσω ένα βράδυ μόνο στη Γάζα και επομένω μπόρεσα τελικά να μείνω, μάλλον δεν μπόρεσα να την νυχτερεύσω, μπόρεσα να μείνω μόνο από τι 9 το πρωί ω τι 3 το μεσημέρι. Αυτό περιορίσε πάρα πολύ το εύρο τελικά τη παρουσία μου εκεί. Θέλαμε πάντως να δούμε πώ αξιοποιούνται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου και προσπάθησα να αξιολογήσω, να αποτιμήσω και να εκτιμήσω τα προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι κυρίως στη Λόριδα της Γάζας και όπως σας είπα είχα και τη δυνατότητα όμως να πάω και στη Δυτική Όχθη. Όσον αφορά το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό τώρα της αποστολής. Βάσει επίσης μιας έκθεσης που συνέταξα και η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μου, πήγα και στην Ισραηλινή πλευρά, στη, στη συνοριακή περιοχή και στην ίδια τη Γάζα και στη δωρεά της Γάζας, στο Κεραίμ Σαλόμ που είναι το πέρασμα αυτό όσον αφορά τα διάφορα προϊόντα, τα εμπορεύματα, όσον αφορά τα τρόφιμα. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση όλα αυτά τα φορτηγά, 800 περίπου φορτηγά φτάνουν στη Γάζα και 80 περίπου, το περιεχόμενο 80 περίπου φορτηγών πηγαίνει προς το Ισραήλ και προ άλλε ε, χώρες. Υπάρχει ένας πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος όσον αφορά τα προϊόντα αυτά. Οι ε, Ισραηλινοί προφανώς ε, δεν θέλουν κανένας εξοπλισμός να βρεθεί στα προϊόντα αυτά, να μην υπάρχει τίποτα το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία όπλων ή για τη διάνοιξη τούνελ ανάμεσα στην Γάζα και το Ισραήλ. Καταλαβαίνετε ότι ε, το όλο πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ αυστηρό, επιβάλλονται πάρα πολλοί περιορισμοί από το Ισραήλ και επομένως η Γάζα έχει καταλήξει να είναι ένα είδος γκέτο. Η ανοικοδόμηση στη Γάζα, όπως φαντάζεστε, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Η οικονομική κατάσταση είναι εντελώς δραματική. Η ανεργία έχει φτάσει το 40% και η ανεργία των νέων είναι 60 περίπου και όλα τα άτομα τα οποία συνομίλησα μου είπανε ότι ε, οι κάτοικοι της Γάζας έχουν την εντύπωση ότι δεν έχουν πλέον μέλλον. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσα να δω ότι υπάρχουν κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες στον ιδιωτικό τομέα, πρωτοβουλίες οι οποίες ξεκινάνε από επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, πήγα σε μια επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας, η οποία ήταν ιδιαίτερα δυναμική η οποία πιστεύει ότι όντω υπάρχει οικονομικό μέλλον για την περιοχή. Πήγα επίση σε μια, περιοχή, σε μια επιχείρηση παραγωγή ρούχων για τα παιδιά και για του νέου, Ρούχα τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και στην περιοχή αλλά και σε διάφορε χώρε τη Ευρώπη. Πήγα επίση σε διάφορα σημαντικά έργα υποδομών, συγκεκριμένα σε ένα εργοστάσιο επεξεργασία λιμάτων, το οποίο εδώ και 10 χρόνια το χτίζανε 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί για τη δημιουργία της μονάδας αυτής επεξεργασίας λιμάτων, αλλά τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί το εργοστάσιο αυτό. απαιτούνται επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ και βλέποντας τις δυνατότητες ε, λειτουργίας ε, του εργοστασίου, του εργοστασίου αυτού, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει κατασκευαστεί όμως όλο το δίκτυο το οποίο θα πρέπει να πλαισιώνει τη μονάδα αυτή προκειμένου πραγματικά τα λιμάτα να καταλήγουν από τις διάφορες κατοικημένες περιοχές προς τη μονάδα αυτή επεξεργασίας των λιμάτων. Και βλέπουμε ότι βρισκόμαστε εκεί 100 μέτρα περίπου από τα Ισραηλινά σύνορα και βλέπουμε εκεί ότι και οι ίδιοι οι αγρότες του Ισραήλ θα ήθελαν να μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό και να μπορούν τα ε, λίμματα τα οποία φεύγουν από το εργοστάσιο αυτό να χρησιμοποιηθούν για την ε, λίπανση των κτημάτων τους. Έχουμε επίσημη πρωτοβουλία της Ούντρα για μικροχρηματοδότηση. Πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική, απευθύνεται πάλι σε ε, μικροεπιχειρηματίες και νομίζω ότι θα μπορούσαμε και εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουμε περισσότερο τέτοιες δραστηριότητες προκειμένου να ενθαρρύνουμε αυτές τις ε, πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι περισσότερα πράγματα μπορούν να γίνουν για την κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση των νέων για τα προγράμματα μαθητείας τα οποία θα μπορούσαν να λάβουν χώρα. Ξέρετε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχουν βέβαια και απαραίτητε επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να λάβουν αυτή την κατάρτιση των νέων. Αυτά όσον αφορά την ε, Δυτική Όχθη. Ήρθα σε επαφή με Βεδουίνους προσπάθησα να καταλάβω τις δικές του συνθήκες ζωής, αυτό, την, αυτή την αναγκαστική εκτόπιση την οποία υφίστανται, επειδή απλώνται όλο και περισσότερο οι επικισμοί του Ισραήλ. Μου ανέφεραν λοιπόν οι Βεδουίνοι τα δεινά στα οποία, στα οποία υφίστανται εξαιτία αυτής της αναγκαστική εκτόπισης. Ξέρετε ότι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία, έχοντας όμως κάποια μικρά κοπάδια με εγωπρόβατα, τα βασικά τους ε, έσοδα προκύπτουν κυρίως από κάποια γεωργική δραστηριότητα στην ε, δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού. Από εκεί πέρα καταφέρουν, ε, δεν ξέρω ακριβώς με ποιες δραστηριότητες, να αποκτήσουν τα απαραίτητα προζωή. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και καταστροφή υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται κυρίως για υποδομές μικρής κλίμακας, και νομίζω ότι μιλάμε περίπου για κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που έχουν χαθεί κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει πολύ αρνητικά τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη ζώνη και που θα μπορούσαν να αποφεληθούν από τις σημαντικές αυτές υποδομές. Ξέρετε ότι Πολλές φορές οι Ισραηλοί αθετούν τα όσα προβλέπονται στη Συμφωνία του Όσλο. Μας λέει η Ισραηλινή πλευρά ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα λεγόμενο master plan, να υπάρχει δηλαδή ένα γενικότερο πρώτερο σχέδιο, πλαίσιο, προκειμένου να υλοποιηθούν στη συνέχεια κάποια έργα υποδομής. Πολλέ φορέ βέβαια, αν η Ισραηλινή πλευρά δεν δώσει μια απάντηση έγκριση ανάμεσα μέσα σε 18 μήνε, η σιγή του αυτή μπορεί τελικά να ισοδυναμεί με αδειοδότηση του έργου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δική τη πλευρά κάνει βέβαια ό,τι μπορεί όσον αφορά τα έργα αυτά υποδομή. Προσπαθεί προφανώ να τηρήσει όλε τι διαδικασίε που προβλέπονται. Αυτό άλλωστε πράττει πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιε περιπτώσει. Και είδα για παράδειγμα ότι έχει δημιουργηθεί ένας δρόμος, μια οδική οδός, ο οποίος δημιουργήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η άσφαλτος έχει στρωθεί όπως πρέπει, έχουν ε, δημιουργηθεί οι, τα παράτητα νησόπεδα επίπεδα προκειμένου να διαχωριστεί ο δρόμος αυτός από τις κατοικίες που βρίσκονται δίπλα. Παρ' όλα αυτά όμως δεξιά και αριστερά από το δρόμο αυτό τελικά δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Ο δρόμος αυτός φτάνει στην είσοδο του χωριού και βλέπουμε ότι εκεί πέρα η υποδομή σταματά. η ασφαλτοποίηση, δεν υπάρχουν φανοστάτες στο χωριό αυτό. Νομίζω ότι θα έπρεπε τα πράγματα να ακολουθούν διαφορετικό δρόμο. Θα ήταν πιο λογικό καταρχάς να υπάρχει απαραίτητη υποδομή μέσα στο ίδιο το χωριό, και να μπορεί τελικά ο δρόμος αυτός, αφού, φτάνει, αφού ολοκληρωθεί, να φτάνει πραγματικά μέσα στο χωριό αυτό. Δεν ξέρω αν τελικά και οι διαδικασίες που ακολουθούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ απαιτητικέ και τελικά δεν προσαρμόζονται πραγματικά στις προσδοκίες και στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Ενδεχομένως να πρέπει να γίνει μια άλλη ιεράρχηση προτεραιοτήτων ή ενδεχομένως να, υπάρχει, ε, να πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος ε, ελιγμός ε, δυνατότητες ελιγμού όσον αφορά την ιεράρχηση αυτή των προτεραιοτήτων. Έπειτα, θα μπορούσα να πω ότι μετά την αποστολή αυτή κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα και κάποιες συστάσεις. Εν γέννη θα έλεγα ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σφαιρική, ένα σφαιρικό όραμα για το τι θέλουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε στην Παλαιστίνη και υπάρχει και μια κάποια έλλειψη συντονισμού. Προφανώς υπάρχει εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόπου. Οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν είμαι όμως βέβαιος ότι πραγματικά τους δίδονται σαφείς οδηγίες, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο οδικός χάρτης. Επίσης εμπλέκονται πολλές και διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά και πάλι έχουμε και εκπροσώπηση από τα ίδια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν έχω πραγματικά την εντύπωση ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο, ιδίως σε σχέση με, τους, ε, με τις υπηρεσίες αναπτυξιακής συνεργασίας των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, δραστηριοποιούνται επί τόπου. Σίγουρα στη Γάζα δεν υπάρχει κυβερνητικό συντονισμό. Η Χαμάς δεν νομίζω ότι ασχολείται καθόλου. Απουσία λοιπόν τέτοιου διοικητικού και τοπικού συντονισμού δεν είμαι πραγματικά πεπισμένο ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να επιτελέσει σωστά το έργο της. Και πραγματικά δεν υπάρχει ένας οργανισμός που να έχει αναλάβει γενικά και σφαιρικά το συντονισμό. Σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που αναφέρθηκα πριν από λίγο του ιδιωτικού τομέα, στον οικονομικό κλάδο, ως προς αυτές νομίζω ότι θα πρέπει να ευνοήσουμε περισσότερο τις δράσεις εκείνες οι οποίες θα συμβάλλουν στην ε, δημιουργία ενός οικονομικού ιστού, να προωθήσουμε περισσότερο τη μικροχρηματοδότηση και τα μικρά αυτά έργα οικονομικά, πολύ περισσότερο από ότι τα μεγάλα οικονομικά έργα, τα οποία πολλές φορές τελικά δεν ολοκληρώνονται ή ακολουθούν διαφορετικό δρόμο από αυτόν που είχαν πάρει στην αρχή όταν πρωτοεγκρίθηκαν. Είδα κάποια έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν με την Μεσόγειο, είδα κάποια έργα που έχουν να κάνουν με την αφαλάτωση των υδάτων. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα μεγαλεπίβολα αυτά έργα. Είναι πολύ σημαντικό η συμβολή μα να είναι τελικά αποτελεσματική θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητε προποθέσει προκειμένου να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Γάζας και Ισραήλ όσον αφορά το πόσιμο νερό και όσον αφορά την επεξεργασία των λιμάτων. Και προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, είναι πολύ σημαντικό, όπως και πριν από 20 χρόνια, και ξέρετε ότι το 1996 είχα πάει στη Γάζα και είχα δει τότε ότι υπήρχαν κάποιες βιομηχανικές μονάδες πάνω στη Μεθόριο μεταξύ Γάζας και Ισραήλ και οι επιχειρήσεις αυτές επέτρεπαν σε πολλούς ανθρώπους που κατοικούσαν στη Γάζα να έχουν μια επαγγελματική δραστηριότητα. Σε ποια συμπεράσματα λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε όσον αφορά το πολιτικότερο επίπεδο. Επ' αυτού, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας πω ότι συμμετέχω στην Επιτροπή Προπολογισμών. Είμαι πρόεδρος στην Επιτροπή Προπολογισμών. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υπερβώ τις αρμοδιότητές μου. Συντοπίω ότι είναι η δική σας η Επιτροπή η πλέον αρμόδια για το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, ποιος μπορούμε να πούμε, να πούμε ότι είναι η έμεση κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Ισραήλ και των υπόλοιπων περιοχών. Και τι κάνει επίσης και η διεθνής κοινότητα, η οποία προσπαθεί να φυσήσει μια κάποια ελπίδα στην Παλαιστίνη, σύμφωνα με τον κοινά θεωρητικά αποδεκτό στόχο για την βιωσιμότητα των δύο πλευρών και του Ισραηλινού κράτους. Αναλαμβάνουμε δράση και στο ανθρωπιστικό πεδίο και νομίζω ότι ε, επ' αυτού το Ισραήλ θα πρέπει να είναι ικανοποιημένο. Ήρθα σε επαφή με τον στρατηγό αυτό που είναι ε, ε, επικεφαλής για τη συνεργασία μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή. Ασχολείται και αυτός πάρα πολύ με το λεγόμενο master plan, το γενικό αυτό σχέδιο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει. Προσπαθεί να εξισορροπήσει στο μέτρο του δυνατού τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αναλάβει ένα ρόλο πολιτικό λίγο πιο έντονο λίγο πιο αναγνωρίσιμο, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια αποσύνδεση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην θέση που έχουμε ως βασικό οικονομικό εταίρο της Παλαιστίνης και το βασικό εταίρο οικονομικό επίσης σε σχέση με το Ισραήλ, ενώ από πολιτικής πλευράς όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει θα έλεγα στο περιθώριο. Η αποσύνδεση λοιπόν αυτή πραγματικά δημιουργεί κάποιες απορίες. Δυσκολεύεται επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με ανοιχτό τρόπο με τους Ισραηλινούς και Παλαιστίνους εταίρους. Είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθεί στο Ισραήλ και να ασκήσει πίεση προκειμένου να μειωθούν οι περιορισμοί που επιβαρύνουν τους Παλαιστίνιους. Ξέρετε ότι οι Παλαιστίνοι προσπαθούν να περάσουν από το ΕΡΕΣ, αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί και νομίζω ότι απομακρύνεται όλο και περισσότερο η προοπτική της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους. Και προφανώς βέβαια θα πρέπει αυτό να λάβει χώρα συνάμα με την προστασία του Ισραήλ από πλευράς ασφάλειας. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς και στις δύο πλευρές. Είναι σημαντικό όμως να μιλήσουμε και με τους Παλαιστινίους, προκειμένου και αυτοί να δεσμευτούν για την εθνική συμφιλίωση και να δείξουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα και διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση των διοικητικών του διαδικασιών, των δημόσιων διαδικασιών του, ιδίω όταν αυτέ έχουν να κάνουν και με χρηματοδότηση που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε και εμεί να παρακολουθούμε ποια είναι η χρήση που γίνεται των ευρωπαϊκών κονδυλίων που χρησιμοποιούνται επί τόπου. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δώσουμε μία προοπτική για ένα κάποιο μέλλον στην Παλαιστίνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι με τους οποίους συνομίλησα και οι οποίοι λένε ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει μέλλον για αυτούς. Να μιλήσουμε λοιπόν και με τις δύο πλευρές προκειμένου να ξεκινήσει εκ νέου διαδικασία, μια διαδικασία που θα πρέπει να ξεπεράσει την στήρα ρητορική, της επαναλήψης που ακούσαμε μετά τη Συμφωνία του Όσλο πριν από 20 χρόνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ πρόεδρε, αυτέ είναι κάποιε παρατηρήσει που θα μπορούσα να κάνω και τις οποίε καταλήγω μετά την αποστολή μου αυτή και τι οποίε έχω τη χαρά να εκθέσω εδώ στη δική σα την Επιτροπή. Και με ιδιαίτερη χαρά θα ακούσω και τι δικέ σα παρατηρήσει. Για άλλη μια φορά, να επαναλάβω ότι απλώ εκπροσωπούσα την Επιτροπή Προπολογισμών, προσπαθώντα καταρχά να δώσω ένα τέλο στα πέντε αυτά χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο μην το ξεχνάμε ότι είναι συνομοθέτη σε δημοσιονομικά ζητήματα, δεν μπορούσε να πάει επί τόπου και είναι ο σημαντικότερος χρηματοοικονομικός εταίρος της Παλαιστίνης. Παραλαμβάνω, δεν μπορούσαν οι ευρωβουλευτές όλα αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια να πάνε στην Παλαιστίνη. Λάβουμε πλέον μια άδεια, μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε επί τόπου και να αποτιμήσουμε πραγματικά τον αντίκτυπο και την επίπτωση των κοινοτικών δράσεων υπέρ των Παλαιστινίων. Ευχαριστώ πολύ, λέγει ο Πρόεδρος. Αγαπητέ συνάδελφε, για αυτή την έκθεση, ο κύριος Καν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Να σας ευχαριστήσω για την αναφορά που μας δώσατε από την επίσκεψή σας. Περιγράφει μια ζωφερή εικόνα η οποία υπάρχει επιτόπου στην περιοχή εκεί και εγώ νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο όταν ζητάτε να υπάρξει περαιτέρω πίεση για μια ειρηνευτική διαδικασία. <clears throat> Αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε ότι υπήρξε τεράστια καταστροφή στην ε, Γάζα. Πόση από αυτή την καταστροφή έχει, από αυτή η καταστροφή έχει αποκατασταθεί. Επίσης, το φως αυτό που είπατε, πώς μπορεί να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα βελτιωθούν οι προοπτικές για, το, για τη Λόριδα της Γάζας. Ποιες είναι οι δυνατότητες να πάει μια αντιπροσωπεία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πάει να δει πιο πολλά πράγματα, γιατί είπατε ότι είχατε πολύ περιορισμένο χρόνο στη Λόριδα της Γάζας. Και τέλος, μια τελευταία παρατήρηση, όταν άκουσα αυτά που είπατε, σκέφτηκα το εξής. για τους πολίτες που ζουν στη Γάζα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να ζει στη Γάζα και του να ζει σε μια ανοιχτή φυλακή. Πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση αυτών των ανθρώπων κατά την άποψή σας. η κυρία Αουκέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω το γεγονός ότι είδατε ότι η Ευρώπη πληρώνει, αλλά δεν έχει κανένα ρόλο στην κατεχόμενη Παλαιστίνη. Και επίσης χαίρομαι που κατανοήσατε ότι οι Παλαιστίνοι είναι άνθρωποι με πολλά ταλέντα και προσόντα, αν τους δώσει κάποιος μια ευκαιρία. Αλλά είναι αδύνατον <clears throat> να εξαγάγει κανείς προϊόντα από τη Γάζα, ακόμα και αν έχει χρήσιμο προϊόντα. Δεν μπορούν να βγουν τα προϊόντα αυτά από τη Γάζα. Το είχα δει στο παρελθόν και τώρα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εγώ είμαι πάρα πολύ απαγοητευμένη και από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε αυτή η επίσκεψη και η παρουσίασή σας. Αυτά δεν ανταποκρίνονται στην εντολή που έδωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε ανταποκρίνονται στις θεμητές μας προσδικίες. Αυτή η επίσκεψη είχε αποφασιστεί τον Ιούνιο του 2015 μετά από πολλές άκρατες προσπάθειες της αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη που να υπάρξει κάποια αντίδραση για, τον, για την άρνηση των Ισραηλινών αρχών να επιτρέψουν την πρόσβαση βουλευτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2011 μέχρι τότε. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους κύριους χορηγούς προς τους Παλαιστάνιου και παρόλα αυτά δεν έχουμε αυτό το βασικό δικαίωμα να επιθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται αυτά τα κονδύλια. Εξάλλου η Γάζα είναι μία από τις πιο ζωφερές και σκοτεινές περιοχές αυτού του κόσμου. <clears throat> Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλοί άλλοι φορείς εξακολουθούν να, να σιωπούν για αυτή την απόλυτα απαράδεκτη κατάσταση. Έγινε δυνατό ο κύριος <clears throat> να συμφωνήσει να υπάρξει μια κοινή δράση από την ΑΦΕΤ και την ΔΕΒΕ και δεσμεύτηκε να γίνει η επίσκεψη αυτή μέσα σε δύο μήνες. Οι δύο μήνε έγιναν 12 Δυστυχώ αλλά είναι ακόμα πιο λυπηρό ότι το αρχικό σχήμα δεν έχει τηρηθεί και έχουμε πάρει μονάχα την δική σας αναφορά. Το μόνο αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης που έγινε πριν από πέντε μήνες, πέντε μήνες ήταν το, η, η εγγραφή, που, το blog που έκανε ο κύριος Αρτουή στην ιστοσελίδα του και μόνο στα γαλλικά. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια επίσημη έκθεση από τον κύριο Αρτουή, η οποία να διανεμηθεί σε όλες τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρχε προβλεπόταν πόροι ανθρώπινη και ηλική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μονάχα για να μονάχα η ιστοσελίδα του κυρίου Αρτουή. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια επίσκεψη και άλλων βουλευτών το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που γυρίσατε ε, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες σώσκια και είχαμε την πρόθεση να πάμε ως αντιπροσωπεία στην Παλαιστίνη πριν από λίγους μήνες και δεν μας επέτρεψε κανένας να πάει στη Γάζα. Η κατάσταση αυτή όπως περιγράφει από την κυρία Άουκεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει. Για να το πω με μεγάλη επίοικια. Είναι μια κατάσταση που δεν έχει τροποποιηθεί εδώ και χρόνια, αν όχι εδώ και δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να βελτιώσει την ε, κατάσταση ζωής των Παλαιστινίων που ζουν στην Ελλάδα της Γάζης. Όταν ακούμε τις φωνές που προέρχονται από το Ισραήλ, συμπεραίνουμε ότι μία λύση δύο κρατών είναι κάτι το οποίο έχει πια, δεν έχει καμιά δυνατότητα επιβίωσης. Δεν είναι μια εφικτή λύση πια, αλλά το <clears throat> δικό μου ερώτημα είναι κάπως διαφορετικό. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη για το λόγο για τον οποίο δεν επιτρέπεται σε κανένα από εμάς να πάει στην Γάζα, στην Λόγια της Γάζα για τα τελευταία πέντε χρόνια χοντρικά, ενώ εσείς μπορέσατε να πάτε δείχνει αυτό μια κάποια αλλαγή πολιτικής από την πλευρά του Ισραήλ. Είναι τύψη συνειδήσεων που έχουν οι Ισραηλοί έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το εξηγείται λοιπόν αυτό το γεγονός, αυτή την έστω και ίσονα αλλαγή αντιμετώπισης από το Ισραήλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτιμώ τις προσωπικές προσπάθειες που ανέλαβε ο κ. Αρτουή για να ταξιδέψει στην Γάζα. Η κατάσταση οπωσδήποτε δεν είναι ικανοποιητική, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να αναφερθούν. Αναφέρατε 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Παλαιστινιακή Αρχή. και νομίζω πως ε, πολλά από αυτά τα λεφτά πάνε για κοινωνικο-οικονομικές υποδομές για να στηρίξει την καθημερινή ζωή των ντόπιων, αλλά έχουν ακουστεί κάποια πράγματα και για απάτη και διαφθορά και παράνομη χρήση αυτών των κονδυλίων για στρατιωτικούς σκοπούς. Ε, για να φτιάξουν, παραδείγματος χάρη, τούνελ ή να αγοράσουν όπλα που χρησιμοποιούνται και πάλι για τρομοκρατικούς σκοπούς. Κύριε Αρτούη, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πηγαίνουν ε, ή καταλήγουν ε, σε νόμιμες χρήσεις. Ευχαριστώ, Σαφχάουζερ. Και εγώ θα ήθελα να κινηθώ προς την ίδια κατεύθυνση. Και εγώ ήμουν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνεργασίας. Είχαμε ένα σχέδιο στη Γάζα που χρειάστηκε να το κλείσουμε. Και εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν προβλήματα με κατάχρηση κονδυλίων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν είσαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούνται σωστά αυτά τα 300 εκατομμύρια που δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, μήπως έχει νόημα να δαπανούμε 300 εκατομμύρια, ίσως θα ήταν καλύτερα να δίνουμε την τεχνογνωσία μας και την ικανότητα που έχουμε να δημιουργήσουμε σχέδια και να προτείνουμε την υλοποίηση αυτών των σχεδιών σε χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι το Κατάρ, όπως είναι κάποιες άλλες χώρες που έχουν πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα και είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τους αδερφούς μουσουλμάνους που έχουν εξουσία στη Γάζα. Θέλω κι εγώ το ερώτημα λοιπόν του πόσο σωστή είναι η δική μας παρέμβαση, μήπως θα έπρεπε αντί να κάνουμε εμεί σχέδια, να τα παρουσιάσουμε σε αυτούς οι οποίοι νιώθουν ότι είναι κοντά σε αυτούς που έχουν εξουσία στη της Γάζας. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Γκόμες. Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να έρθω προηγουμένω και να ακούσω αυτά που είπε ο κύριο Σαρτούη. Θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα μετά από αυτά που είπε και η συναδελφή μου. Κάποτε κάποιο Τόνι Μπλερ είχε οριστεί ω εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Λεωρίδα τη Γάζας. Και υπήρχε και ένα σχέδιο αποχέτευσης και διαμαρτυρόταν ότι δεν μπορούσε να πετύχει να προχωρήσει αυτό το σχέδιο γιατί υπήρχαν κάθε είδους πολιτικά εμπόδια. Η Γάζα είναι πραγματικά μια ανοιχτή φυλακή. Ήτανε όταν πήγα και τώρα πρέπει να είναι ακόμα χειρότερη. Αυτό το οποίο πραγματικά με ενόχλησε είναι ότι αυτή ήταν μια σαφής περίπτωση που εμείς πληρώναμε αλλά δεν μετρούσε ο λόγος μας. Και φαντάζομαι ότι η κατάσταση αυτή έχει γίνει ακόμα χειρότερη. Δεν είναι το θέμα που τα χρήματα πώς, πώς χρησιμοποιούνται. Όταν δίνουμε χρήματα στην ούνρα, πάντα τα χρήματα αυτά φτάνουν στους αποδέκτες Το ερώτημα είναι, αν δεν υπάρξει καμία κίνηση για να ξαναρχίσουν οι, οι νευτικές ε, διαδικασίες, έχει νόημα εμείς να χρηματοδοτούμε αυτή την ανοιχτή φυλακή, γιατί αυτό κάνουμε τελικά. Κύριε Πρόεδρε, από Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω βέβαια αν είμαι σε θέση να απαντήσω σε ερωτήσεις αυτές. Και λυπάμαι, λυπάμαι πραγματικά να η συμμετοχή μου στην αποστολή αυτή δημιουργεί αυτή τη στιγμή ερωτηματικά ή αν έχει απογοητεύσει τελικά κάποιους. Αυτό το οποίο πρέπει να θυμηθούμε είναι το εξή. Από τότε που πήρε την εξουσία η Χαμά στη δουλειά τη Γάζας, το 2006 δηλαδή, και από τότε που ε, το Ισραήλ επέβαλε αποκλεισμό, το 2007, οποιαδήποτε επίσκεψη στη δουλειά τη Γάζας υπόκειτο σε μια αδειοδότηση από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Και Υπήρχαν πάρα πολλές απογορεύσεις για λόγους ασφάλειας και αυτό το λόγο δεν καταφέραμε εμείς από το 2011 και μετά να κάνουμε καμία επίσημη αποστολή επιτόπου. Η κατάσταση όμως έκτοτε εξελίχθηκε και στο νέο αυτό λοιπόν πλαίσιο ο πρόεδρος Σούλτς ενημέρωσε τον πρόεδρο της Επιτροπής ΑΦΕΤ, την πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και ήρθε σε επαφή και εμένα τον ίδιο και είπε το 2005 ότι θα ήταν πλέον σκόπιμο να πάμε στη όρθα της Γάζας για μία πρώτη επίσκεψη και να ανοίξει κατά κάποιο τρόπο πάλι η δυνατότητα αυτή να επισκεπτόμαστε την περιοχή. Όπως σας είπα ήταν πολύ δύσκολο να συμπέσουμε με τον κύριο Μπρόκο και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να πάω μόνος. Και σας είπα στη συνέχεια τι είδα επί τόπου. Επαναλαμβάνω σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ να υπερβώ τι αρμοδιότητέ μου. Πήγα εκεί ω πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμών. Και όταν πηγαίνει κανεί μόνο για 24 ώρε, προφανώ δεν μπορεί να κάνει διεξοδικό έλεγχο, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούσα πραγματικά να δω ότι όντω τα τιμολόγια ανταποκρίνονται πραγματικά στα χρήματα τα οποία δώσαμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο τελικό προϊόν. Αναγκαστικά έπρεπε να μείνω λίγο στην επιφάνεια των πραγμάτων. Ήθελα να επισκεφθώ κάποιε μονάδε, κάποια κέντρα, να επισκεφθώ κάποιε επιχειρήσει να πάω σε μια συνάντηση που είχε οργανώσει η Ούνρα, ένα μικρό, μια μικρή τοπική έκθεση στην οποία συμμετείχαν παραγωγοί οι οποίοι είχαν χρηματοδοτηθεί από τη μικροχρηματοδότηση της Ούνρα, αλλά και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Δεν είμαστε οι μόνοι προφανώς που χρηματοδοτούμε επιτόπου. Δεν μπόρεσα λοιπόν να αποκρισταλώσω μια τελική άποψη, το καταλαβαίνετε αυτό, είναι απόλυτα λογικό. Και ο πρώτος συνάδελφος που πήρε το λόγο μετά την παρέμβασή μου, με ρώτησε αν τελικά πρόκειται για μια ανοιχτή φυλακή. Εγώ σας είπα, χαρακτήρισα την ορίδα της Γάζας ένα γκέτο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κανείς από το γκέτο αυτό. Και τα προϊόντα περνάνε από το μόνο σημείο διέλευση στο Κερέν Σαλόμα, είναι προϊόντα τα οποία περνάνε από εξονυχιστικό έλεγχο. Γιατί ε, οι Ισραηλινοί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε προϊόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του Ισραήλ. Και δεν έπρεπε κανείς ε, να περάσει από το σημείο αυτό ούτε καν υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την διάνοιξη σειράγκων μεταξύ της δωρίδας της Γάζας και του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ένταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχουν πάρα πολλές ε, υποψίες και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επιζήμιες συνέπειες. Είδα ότι υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια κτίρια που βρίσκονται σε πολύ δεινή κατάσταση, είδα πραγματικά τις επιπτώσεις του πολέμου και είδα ότι όντως ακόμα και τα έργα καθυστερούν πάρα πολύ γιατί δεν υπάρχει ο παρέτος συντονισμός. Υποτίθεται ότι οι δημοτικές εκλογές θα γινόντουσαν τον Οκτώβριο. Σε αυτές ε, υπολόγιζαν πάρα πολλοί τοπικοί παράγοντες προκειμένου να υπάρχει τελικά ένα συντονιστικό φορέας και είμαστε ήδη μέσα Νοεμβρίου και δεν έχει συμβεί τίποτα. Στο Κέρεν Σαλόμ, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Αιγυπτό, πραγματικά μπορούσα να δω ποιε ήταν οι επιπτώσεις και στο ίδιο το Σινάι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα σταθές, η ασφάλεια είναι πολύ σχετική, πολύ επισφαλής. Το πέρασμα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου ήταν κλειστό επίσης. Και όσον αφορά την κυρία Όγκεν, η οποία είναι αντιπρόεδρος της ε, Αντιπροσωπείας των Σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παλαιστίνης, πρέπει να σας πω ότι με κάλεσε η αντιπροσωπεία σας τον Οκτώβριο. Ελπίζω πραγματικά να διασκεδάσω κατά κάποιο τρόπο την απογοήτευση αυτή που σας προκάλεσε η έκθεση μου αυτή. Όπως σας είπα, ως ε, Ευρωβουλευτής έπρεπε στη συνέχεια να καταγράψω τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής, να δω αν θα μπορούσα να αντλήσω κάποια διδάγματα και να προσπαθήσω να καταλήξω και σε κάποιες συστάσεις. Αυτό προσπάθησα στεκα να κάνω. Κανονικά θα ερχόμουν εδώ πέρα το Δεκέμβριο και προφανώς ε, θέλω να έρθω και σε επόμενες συνεδριάσεις ε, της Επιτροπής σας και είχα προτείνει μάλιστα στο παρελθόν το 2017 να γίνει μια, ε, επίσκεψη στο Ιδρά της Γάζας ως συνέχεια της δικής μου της αποστολής. και στην επίσκεψη αυτή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στα μέρη τα οποία θα μπορούσαμε να επισκεφθούμε. Λυπάμαι επίσης που η έκθεση αυτή ε, συνετάχθη μόνο στα γαλλικά, αλλά προφανώς μπορεί να μεταφραστεί η έκθεση αυτή προκειμένου όσοι θέλουν να τη διαβάσουν προκειμένου όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το διδαπιτόπου να το πράξουν. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να πετύχω τίποτα παραπάνω με την έκθεση αυτή πέρα από το να καταγράψω τα όσα έζησε επιτόπου. Όπως σας είπα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επιβάλλει πολύ συγκεκριμένου κανόνες σύμφωνα με τους οποίους δεν μπορούμε να διανυκτερεύσουμε επιτόπου. Εγώ τουλάχιστον σε επικεφαλής αποστολής δεν μπορούσα να διανυκτερεύσω στην πλευρά της Γάζας. Μόνο ορισμένοι μόνο συμμετέχονται σε συγκεκριμένε αποστολέ μπορούν να διενυκτερεύσουν. Το βρίσκω αυτό πολύ περίεργο γιατί ο κανόνα αυτό δεν επιβάλλεται από τι εθνικέ αντιπροσωπείε των κρατών μελών παρά μόνο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Επαναλαμβάνω πάντω ότι στα πλαίσια τη έκθεσή μου αυτή προσπάθησα να κάνω ένα απολογισμό, να καταλήξω απλώ σε κάποια συμπεράσματα και σε κάποιε συστάσει. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα των πραγμάτων, αν και εμείς έχουμε ένα πιο ξεκάθαρο όραμα για το τι θέλουμε να κάνουμε στην Παλαιστίνη, ήρθα σε επαφή, σε επαφή με εκπροσώπου των πολιτών επιτόπου και πραγματικά έθεσαν το ζήτημα αυτό, το ότι δεν υπάρχει ο δικός χάρτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουμε θέσει προτεραιότητες, για ποιο το λόγο ευνοούμε τη μία διαδικασία εις βάρος της άλλης. Αναφέρθηκα πριν από λίγο στο παράδειγμα εκείνου του δρόμου που έχει κατασκευαστεί μένα αλλά δεν φτάνει τελικά μέσα στο χωριό. Έχουμε ακολουθήσει για το έργο αυτό συγκεκριμένα τους κανόνες που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση έργων υποδομής, αλλά δεν νομίζω ότι τελικά ευνοούμε τα πραγματικά συμφέροντα των πολιτών, τη στιγμή που ο δρόμος δεν φτάνει καν μέσα στο χωριό. Όπως σας είπα επίσης και απαντώ και σε άλλες ερωτήσεις, προσπάθησα να κάνω ένα πρώτο βήμα, να βγούμε από το διέξοδο αυτό στο οποίο βρισκόμασταν, από το ότι δεν μπορούσαμε εδώ και πέντε χρόνια να πάμε στην Παλαιστίνη, μολονότι είμαστε ο πιο σημαντικός χρηματοδότης της περιοχής, μια κατάσταση που ήταν σαφώς απαράδεκτη. Με ρωτήσατε αν είμαστε πραγματικά σίγουροι και πεπισμένοι ότι τα όσα χρηματοδοτούμε δεν αποτελούν αντικείμενο διασπάθησης ε, χρημάτων ή παρατυπιών. Πραγματικά δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή οριστικά για το ζήτημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί με διαγωνισμούς. Υποτίθεται ότι εμπιστεύεται τοπικές επιχειρήσεις και θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά προσεκτικό σε αυτά που θα πω, αλλά στα πλαίσια της ανθρωπιστικής δράσης που χρηματοδοτούμε και σε άλλες περιοχές, πραγματικά δεν είμαι πεπισμένο ότι ένα μέρος των χρημάτων πραγματικά πηγαίνει σε όλου, τους σωστού αποδέκτες και ότι δεν υπάρχει τελικά και ένα τμήμα της χρηματοδότησης το οποίο παίρνει κάποιον άλλο δρόμο ή τελικά αποτελεί αντικείμενο διασπάθησης ή κατάχρησης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ταπεινόθρονες Γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για, για τη χρηματοδότηση άλλων ανθρωπιστικών δράσεων σε άλλες περιοχές του κόσμου. Διασπάθηση χρημάτων, κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θέλω να ελπίζω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έκανα σε καμία περίπτωση εξοχιστικό έλεγχο και επομένω δεν μπορώ να τοποθετηθώ οριστικά. Δεν έκανα λογιστικό έλεγχο δεν κοίταξα τα βιβλία όλων αυτών των επιχειρήσεων. Πήγα σε ένα κέντρο κατάρτισης για απομονωμένες γυναίκες. Ένα σχέδιο το οποίο υποστηρίζει μια μη κυβερνητική οργάνωση. Και φαντάζομαι ότι ε, το αποτέλεσμα, αν θέλετε, είναι θετικό. Το αν κάτι διάρκεια της δημιουργίας του προγράμματο αυτού κατάρτιση υπήρχε διασπάθηση χρημάτων. Δεν το γνωρίζω αν υπήρχαν κάποιε παρατυπίε. Πήγα επίση ε, σε μια γαλακτοκομική βιομηχανία. Πάλι μπόρεσα να δω ότι υπάρχουν αγελάδε και ότι όντω παράγονται προϊόντα, αλλά δεν έλεγξα τα λογιστικά βιβλία τη μονάδα αυτή. Όπω σα είπα, πήγα και στην εργοστάσιο παραγωγή ε, ρούχων για παιδιά που απασχολεί πολλούς ανθρώπους και πραγματικά κάνει μια εξαιρετική εργασία και μάλιστα τα προϊόντα αυτά εξάγονται στο εξωτερικό, αλλά και πάλι δεν μπορούσα να κάνω εκεί πέρα οικονομικό έλεγχο. Από το πέρασμα αυτό που σας είπα, στο σημείο ελέγχου φτάνουν 800 φορτηγά και βγαίνουν μόνο, περνάνε μόνο 80 από την άλλη πλευρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι μπαίνει και τι βγαίνει. Ο Τόνι Μπλερ τώρα. Όντω, αναφερθήκατε κύριε Γκόμε σε αυτή τη μονάδα επεξεργασία λιμάτων. 100 εκατομμύρια έχει στοιχήσει και δεν λειτουργεί ακόμα. Όντω, αυτή τη στιγμή για να φτάσει κανείς στο εργοστάσιο αυτό υπάρχουν πολύ ωραία μαρμάρινα σκαλοπάτια. Δεν λειτουργεί όμω η μονάδα αυτή. Χρειάζονται ακόμα 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ για να αρχίσει να λειτουργεί αυτή η μονάδα επεξεργασία λιμάτων. Δεν είμαι όμω πεπισμένο ότι υπάρχουν και απαραίτητοι αγωγοί προκειμένου να φτάνουν τα λίματα από τι γύρω περιοχέ σε αυτή τη μονάδα επεξεργασία λιμάτων και νομίζω ότι θα έπρεπε, όπως σας είπα, να υπάρχει και μια συμφωνία συνεργασίας με τους αγρότες από το Ισραήλ, οι οποίοι βρίσκονται από την άλλη πλευρά των συνόρων και οι οποίοι χρειάζονται τα λίματα αυτά ως λίπασμα για τα αγροκτήματά τους. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να ξαναδούμε λίγο αυτές τις ε, συμφωνίες ε, που υφίστανται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, όχι μόνο για τα ύδατα, αλλά και για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, για το πόσιμο νερό. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούμε μονάδες αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού και πάλι εδώ πέρα όμως τα αποτελέσματα δεν είναι διασφαλισμένα και από την άλλη δαπανώνται τεράστια ποσά. Μήπως θα ήταν πιο χρήσιμο να προωθήσουμε περισσότερο τη μικροχρηματοδότηση και να χρηματοδοτήσουμε έργα μεσαίας ή μικρής, αν θέλετε, οικονομικής κλίμακας, προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργεία της τάξης 40% στους ανήλικες και 60% στους νέους. Και πάλι, σε ό,τι αφορά την ευτική διαδικασία, αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο κύριος χρηματοδότης, δεν συμμετέχει στι βασικές διαπραγματεύσεις. Εγώ κάθε φορά που υπάρχει ένα σημαντικό γεγονό ψάχνω να δω αν υπήρχε κάποιο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό σα λέω ότι ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψή μου, αλλά ήταν ιδιαίτερα επιφανειακή, γιατί ήταν και σύντομη. Γιατί ήμουνα μόνο. Αλλά φυσικά χρειάστηκε μια περαιτέρω επίσκεψη και αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε το 2017 και αργότερα αλλά σας λέω ποια είναι τα δικά μου συναισθήματα και από άλλες επισκέψεις που έκανα στο Λίβανο, στην Ιορδανία, στην Τουρκία. Νομίζω ότι η τοπική μας εκπροσώπηση δεν νομίζω ότι πάντα ακολουθεί τον οδικό χάρτη που έχει διατυπωθεί με τρόπο χωρίς αμφισημίας. Ναι, βεβαίως θέλουμε κονδύλια, αλλά ποια είναι και η κοινή αντιμετώπιση ποια είναι η κοινή στρατηγική. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει η Επιτροπή ΑΦΕΤ να επιληφθεί για αυτού του ερωτήματος για να δώσει και μια απάντηση. Ο κύριος Μπέλτερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αρτουή για αυτά τα οποία μας είπατε. Ε, θα ήθελα να μάθω τι γίνεται εκεί πέρα με την χριστιανική ε, μειονότητα στην Γάζα. Ε, βεβαίως το θέμα είναι αν υπάρχει κάποια ειδική ε, αντιμετώπιση, αν λαμβάνεται υπόψη η πολύ επισφαλής θέση της χριστιανικής μειονότητας. Αν υπάρχει κάποια στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Υπάρχουν, υπάρχει ένας γνωστός γυναικολόγος ο οποίος δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του μόνο και μόνο γιατί είναι χριστιανός. Καταλαβαίνω πάντω το ερώτημά σα, αλλά στι 24 αυτέ ώρε που πέρασα στη ώρα τη Γάζα και στι επαφέ που είχα επιτόπου, δεν έχω συλλέξει στοιχεία που θα με επέτρεπα να δώσω οριστική απάντηση στο ερώτημά σα. Προφανώ εμπιστευόμαστε τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που δραστηριοποιούνται επιτόπου, οι οποίε θεωρώ ότι δραστηριοποιούνται χωρί διακριτική μεταχείριση αμερόληπτα δεν έχω όμω απαραίτητα στοιχεία αυτή τη στιγμή να σα δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση. Πραγματικά θεωρώ ότι οι δικέ μας απαντήσεις από την ΕΚΟ συγκεκριμένα ακούνε όλες αυτές τις προσδοκίε των πολιτών και ότι βρίσκονται υπεράνω οποιασδήποτε διακριτική μεταχείρισης και σαφώς δεν θέλουν να δημιουργήσουν γκέτο μέσα στον γκέτο. Yeah, just, uh, Mr. Uh- η κυρία Άουκεν, μια παρατήρηση μοναχά. Λοιπόν, δεν θέλω να σταθώ στις δικές μου ερωτήσεις. Θα ήθελα να ακούσω και κάποια σχόλια από την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που είναι παρούσες εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τα δικά του σχόλια για αυτή την έκθεση. Bonjour. Ε, Fuentes. Είμαι από την Υπηρεσία Εξωτερικών ε, Εξωτερικής Δράσης και οι αρμοδιότητες μου έχουν να κάνουν μονάχα με το Ισραήλ και τη διαδικασία ειρήνευσης. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρτουής για την επίσκεψη που έκανε. Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη για μας έχει καλύψει αυτό το κενό το που δημιουργήθηκε επί πέντε χρόνια όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να πάει στη Γάζα. Εμεί ακούσαμε μεγάλη προσοχή και είχα την ευκαιρία να συναντήσω και τον κύριο Αρτούι πριν από το ταξίδι του εκεί. <clears throat> Πήρα ε, και τις, ε, άκουσα και τις απόψεις του και μετά από το ταξίδι. Νομίζω ότι αυτά που μας είπε είναι απόλυτα σχετικά και εύστοχα. Αν έχετε τώρα ένα συγκεκριμένο ερώτημα να μας θέσετε, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Ja, alles gesagt, nur nichts zum Inhalt. Ist das nicht verständlich, wie ich mich ausdrücke? Κύριε Πρόεδρε, αν καταλαβαίνω καλά, η επίσκεψη του Προέδρου Αρτούι είναι μετά από εντολή του Προέδρου Σούλτς, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, συνεργάστηκε για την προετοιμασία αυτής της επίσκεψης και πήραμε και την έκθεση του κυρίου Αρτουής, την οποία αναδυθήσαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μα ποια είναι η κατάσταση κατά την άποψή σας, λέει ο πρόεδρος ε, Μπροκ. Μήπως μπορείτε να μας εκφράσετε τη θέση σας για την κατάσταση, πώς βλέπετε την κατάσταση εκεί. Είναι σωστά αυτά που είπε ο κύριο Ρόγκ, είναι λαθασμένα. Τι θα έπρεπε να κάνουμε, θα έπρεπε, πού θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, που υπάρχουν προβλήματα για την εφαρμογή του προγράμματος. Τι έχετε να πείτε για αυτά. Κατά την άποψή μας, το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε <clears throat> στο Ισραήλ και στις σχέσεις με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη είναι ότι, ότι με τα προγράμματα ανάπτυξης, τα ανθρωπιστικά προγράμματα μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που είναι ενάντια με την προσέγγιση μας. Είμαστε κατά της κατοχής αυτών των εδαφών και στην περίπτωση της Γάζας είμαστε εναντίον του αποκλεισμού της Λόριδας της Γάζας. Καταρχήν δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη που μπορούμε να δώσουμε η οποία να άρει το κόστος της κατοχής. Δεύτερον, όταν θέλουμε να αναπτύξουμε προγράμματα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολιτική κατάσταση η οποία αντιβαίνει στις δικές μας πολιτικές θέσεις. Προσπαθούμε να πείσουμε το Ισραήλ ώστε τα προγράμματα αυτά να αποδώσουν καρπούς. Παραδείγματο χάρη. Ο πρόεδρος Σαρτουή αναφέρθηκε στο σχέδιο αποχέτευσης, στο σχέδιο επεξεργασίας λιμάτων. Έχουμε κάνει επανειλημμένα διαβήματα προς τους Ισραηλούς για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό. Η τελευταία μας επαφή έγινε τον προηγούμενο Σεπτέμβρη και υπήρξε μια συμβιβαστική λύση με το Ισραήλ ώστε να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να λειτουργήσει αυτό το σχέδιο. Επίσης για το σχέδιο αφαλάτωσης και εκεί συνεργαζόμαστε με τους <clears throat> Ισραηλούς και τους Παλαιστίνιους ομολόγους μας για να λειτουργήσει αυτό. Μια δεύτερη γραμμή δράσης από τη δική μας πλευρά. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους Παλαιστίνιους, να δημιουργήσουμε θεσμούς, να τους αναπτύξουμε την ικανότητά τους, ώστε να μπορούμε να, να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα κονδύλια που τους δίνουμε και τρίτον προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κατά γράμμα τους μηχανισμούς δημοσιονομικού ελέγχου που προέρχονται από το ελεκτικό συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε τα κονδύλια μας να μην διασπαθίζονται. Αυτά κάνουμε. Αν η κατάσταση είναι αυτή που θα θέλαμε, φυσικά όχι. Αλλά είναι αυτή που είναι και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε τα κονδύλια μας κάτω από αυτές τις συνθήκες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρόσθετο ερώτημα. Μίλησατε για κατοχή. Οι Ισραηλοί δεν είναι στη δύναμη κατοχή στη Γάζα από ό,τι ξέρω, αλλά μιλάτε για κατοχή από τη Χαμάς. Πώς βλέπετε τη συνεργασία μεταξύ Χαμάς και Παλαιστινιακής Αρχής και αν αυτή ε, βοηθάει ή εμποδίζει την ε, εφαρμογή αυτών των σχεδίων γιατί η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει καμία εξουσία και καμία λειτουργική δυνατότητα να επηρεάσει τα πράγματα στη Γαζή Δεν είναι πρόβλημα αυτό κατά την άποψή σα. Κύριε Πρόεδρε, όταν αναφέρθηκα στην ε, κατοχή εννοούσα την ε, Δυτική Όχθη που ήταν και αντικείμενο της επίσκεψης του Πρόεδρου του. Προφανώς στην Γάζα το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αποκλεισμός για την συνεργασία μεταξύ Χαμάς και Παλαιστινιακής Αρχής. Οπωσδήποτε, εδώ και καιρό ζητάμε την συμφιλίωση των Παλαιστινίων. Η τρέχουσα κατάσταση στην Γάζα δεν βοηθάει, αλλά δεν έχουμε παφές ε, και σχέσεις ε, με την Χαμάς. Αυτό το ακολουθούμε κατά γράμμα και προσπαθούμε να επηρεάσουμε στο μέτρο του δυνατού την Παλαιστινιακή Αρχή στα όσα μπορούν να κάνουν, γιατί έχει πολλούς υπουργού που είναι αρμόδιοι για διάφορα ζητήματα στη Γάζα. Ειδικά για κάποια θέματα υποδομών και η σχέση μας με την Παλαιστινιακή Αρχή ε, αρκεί νομίζω για να έχουν νόημα αυτά τα πράγματα. Συνεργαζόμαστε και με την Ούνρα που έχει διάφορα προγράμματα και στηρίζει τους ε, Παλαιστίνιους στην Γάζα, παρέχει βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση κτλ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Πρέπει να επανέλθω στο ερώτημα που έθεσε ο Μπάς Μπέλτερ. Μπορώ να κατανοήσω ότι έχουμε την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το θέμα το οποίο είναι θέμα προτεραιότητας, ότι υπάρχει μια κοινότητα, μια ομάδα του πληθυσμού η οποία βρίσκεται σε δίωξη, οι χριστιανοί που καταπιέζονται από τη Χαμάς. Και ξέρουμε ότι η Χαμάς είναι ένα πολιτικό σχήμα το οποίο κυβερνά τη Λόγια της Γάζας, ανεξάρτητα από την ιστορία της. Θα πρέπει να εξετάσουμε και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την εξουσία της Χάμας. Της Χαμάς. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός, ασκεί την εξουσία εκεί και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Και τρίτον, θα πρέπει να σκεφτούμε και την ομάδα του πληθυσμού που είναι αντικείμενο διακρίσεων. Το να τους βοηθήσουμε αυτούς δεν σημαίνει διάκριση εναντίον της κοινότητας που ασκεί τις διακρίσεις. Αυτό για να διευκρινίσω ότι κατανοώ από αυτά που είπατε για τις διακρίσεις. Η κυρία Γκόμες. Και εγώ έχω κάποιο ερώτημα. Επί τη βάση αυτού που είδα εγώ η ίδια στη Λόιδα της Γάζας στο παρελθόν, όλοι αντιμετωπίζουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι, οι χριστιανοί, οι άθεοι, όλοι. Γιατί βρίσκονται σε ένα έδαφος όπου δεν υπάρχει κανένα σεβασμός για τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Και δεν ήταν αντικείμενο σεβασμού τα ανθρώπινα δικαιώματα στο παρελθόν γιατί υπήρχε η κατοχή από το Ισραήλ και τώρα γιατί υπάρχει αποκλεισμό από το Ισραήλ. Το ερώτημά μου προς την Κομισιόν είναι εμείς πληρώνουμε την ύφη αυτού του αποκλεισμού. Εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε για να υπάρχει αυτός ο αποκλεισμό. Το Ισραήλ θα έπρεπε να πληρώνει τουλάχιστον να τρώνε αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την ανοιχτή φυλακή ή όχι. Αυτό είναι μια ερώτηση μάλλον προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά αν θέλει και η Κομισιόν να παρέμβει, ευχαριστώ. Αλλά η αποσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λόριδα της Γάζας έχει να κάνει και με τη Χαμάς και όχι μονάχα με το Ζαΐρ. Και η Χαμάς παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, Γάζα. Χωρίς μικρόφωνο κυρία Γκόμες. Αν θέλετε να δώσετε μια σύντομη απάντηση και μετά πρέπει να κλείσουμε να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για το ερώτημά σας και να δώσω μια σύντομη απάντηση. Υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα που πρέπει να τα θέτουμε στον εαυτό μας. Θα ήταν καλύτερα να σταματήσουμε τη συνεργασία, θα βοηθούσε περισσότερο τους Παλαιστινίους. Η απάντηση στην οποία έχουμε καταλήξει μέχρι τώρα είναι όχι. Πιστεύουμε ότι τα προγράμματά μας είναι κρίσιμα για να δημιουργήσουν τις συνθήκε και τις ικανότητε για να είναι βιώσιμο το Παλαιστινιακό κράτος όταν δημιουργηθεί. Βοηθάμε πολλού Παλαιστίνιους, δίνουμε τη δυνατότητα παιδεία, καλύπτουμε τις υγειονομικέ του ανάγκες. Τα προγράμματα μας μπορεί να μην είναι απόλυτα αποτελεσματικά, αλλά καλύπτουν ένα χάσμα το οποίο αλλιώ θα παρέμενε και σίγουρα δεν θα το κάλυπτε ο αραβικός κόσμος που υποστηρίζει την Παλαιστίνη, αλλά δεν έχουν δώσει τα ποσά τα οποία υποσχέθηκαν. Αν δεν είμαστε εμεί, δεν έκανε κανένα τίποτα κατά πάσα πιθανότητα. Ο κ. Σαρτουή για να κλείσει τη συζήτηση. Ακούστε. Μην βάζετε στο στόμα μου πράγματα τα οποία δεν ήθελα εγώ να, να τα πω. Πήγα σε μια σύντομη αποστολή στη Γάζα ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών για να προσπαθήσω να σχηματίσω μια εικόνα για την τοπική κατάσταση και ιδίω ιδίως για τη χρήση των κονδυλίων που τίθενται στη διάθεση της Παλαιστίνης από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Σας παρουσίασα τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά μου. Σας είπα ότι είναι το η Γάζα. <clears throat> η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Αλλά όταν έχετε 40% συνολική ανεργία και 60% ανεργία των νέων, θα πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η προτεραιότητα. Είναι φανερό ότι για μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της συντονισμού και ελείπει κάποιος ο οποίος θα συντονίσει όλη αυτή την αρρωγή που δίδεται επιτόπου <clears throat> στην ε, Γάζα. Ξέρω ότι η Παλαιστινιακή Αρχή σκέφτεται να κάνει κάποιο περιφερειακό σχήμα, ένα σχήμα αποκέντρωση για να είναι ενιαία περιοχή η Γάζα και όταν πήγα εκεί τον Ιούλιο υπήρχαν πολλές προσδοκίες από τις δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο για να δημιουργηθεί μια τοπική εξουσία η οποία θα λάμβανε περισσότερο το γενικό συμφέρον και την κάπως ομαλοποιημένη κατάσταση με το Ισραήλ. Δυστυχώς δεν υπήρξαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και οι Ισραηλινές αρχές αποφάσισαν να αναβάλουν τις εκλογές γιατί θα, θα μπορούσαν να επαληθευτούν στην ε, Λόριδα της Γάζας και θα μπορούσαν να αντικείμενο αμφισβήτηση στα εδάφη της ε, Δυτικής Όχθης. Λοιπόν, τώρα για το αν υπάρχουν κοινότητε οι οποίε είναι υπό δίωξη, ε, σε καταδίωξη, εγώ δεν μπόρεσα να σχηματίσω εικόνα για αυτά τα θέματα και νομίζω ότι ως μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων εσείς είσαστε πολύ πιο γνώστες της κατάστασης από μένα για να εκτιμήσετε κάτι τέτοιο. Αλλά για να μπορέσει να αναθερμανθεί η οικονομία εκεί και αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει με όλα αυτά τα μικροσχέδια που πιστεύω ότι δίνουν κάποια ελπίδα γιατί για μένα το πιο σημαντικό ήταν η άποψη που είχαν οι κάτοικοι της Γάζας ότι δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτούς. Του τουλεχθέντος λοιπόν, ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό προσπάθησα να εξηγήσω, είναι ότι όταν είμαστε ο πρώτος χρηματοδότης σε μια περιοχή, κάποτε θα πρέπει να βρούμε και την σωστή γλώσσα, ώστε να κατανοήσουν οι Ισραηλινές αρχές και οι Παλαιστινιακές αρχές ότι, μα είναι αλήθεια, το είπε και η κυρία Γκόμες, η ανθρωπιστική βοήθεια που δίνουμε εμείς ίσως είναι μια ανακούφιση για το Ισραήλ. Εγώ συνάντησα τον ε, αντιστράτηγο Γιόρντε Χάι, ο οποίος είναι αρμόδιος για την ε, δομή συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, πιστεύει ότι μπορεί να προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση για να ειρηνεύσει η κατάσταση για να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για τους πολίτες της Γάζας. Θα ξανά έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και εγώ θα βρω τρόπο να μεταφράσω στα αγγλικά την εκθεσή μου η οποία δημιούργησε το ενδιαφέρον της Αντιπροέδρου της ε, Αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη. Θα, προσθέσω, λοιπόν, θα προσπαθήσω λοιπόν να συμβάλλω επί τη βάση αυτό που είδα και άκουσα. <clears throat> Είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά όταν είμαστε τόσο σημαντικοί χρηματοδότες, ίσως θα πρέπει να έχουμε και μια πολιτική στρατηγική και ένα πολιτικό όραμα και αυτό πρέπει να το κάνει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ και για την ευγενή πρόσκλησή σας κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση βλέπετε ότι ανακοίνησε το ενδιαφέρον για το θέμα, όπως ε, επίσης και η παρατήρηση της Κομισιόν ανέδειξε την ανάγκη να εμβαθύνουμε στο θέμα. Θα ταξιδέψουμε ούτως ή άλλως στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα και θα παρακολουθήσουμε το θέμα. Και να προσπαθήσουμε και με τα λεφτά που δίνουμε να έχουμε μια καλή επίδραση στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, να βοηθήσουμε κάπως. για να υπάρξει, όπως είπαμε βεβαίως πάνω απ' όλα μια σωστή ε, χρησιμοποίησή τους και να μην πάνε σε λάθος χέρια. Και υπάρχουν πραγματικά περιορισμένες δυνατότητες ε, της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας λόγω ακριβώς ε, της ε, Χαμάς. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ.